Συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Έχετε στέθηση στα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Υπάρχουν σχόλια. Εάν όχι εγκρίνονται τα πρακτικά. Και προχωρώ στο πρώτο θέμα στην ημερήση διάταξη, την έκθεση του κυρίου Φέρμ. Οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας καλωσορίσω και τον κύριο Χόιερ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τον κύριο Μαστρογιάννη, ο οποίος νομίζω είναι εδώ για πρώτη φορά. Ο κύριος Μαυρογιάννης, για πρώτη φορά εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας. Ο κύριος Φέρμα έχει το λόγο. Ε, πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο τίτλος ε, αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα αλλά κρύβει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Είναι τα ομόλογα έργου. Το μέλλον, το οικονομικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σχετίζεται μόνο με την κρίση. Σχετίζεται και με μια πιο μακροπρόθεσμη ε, διατήρηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και συνδέεται με την αύξηση των επενδύσεων που βαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να συνεργαστούμε και ε, να βοηθήσουμε όλα τα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν μεταξύ τους για να εκμεταλλευτούν το δυναμικό τους. Έχουμε 500 εκατομμύρια πολίτες, καταναλωτές την ίδια αγορά. Συνεπώς πρέπει να επενδύσουμε σε σύγχρονες υποδομές στον τομέα της ενέργειας, ε, των μεταφορών και της ψηφιακή εποχή. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε ευφυή ανάπτυξη για όλους. Η οικονομική κρίση δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα της κατάρρευσης του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα. Είναι επίσης αποτέλεσμα του γεγονότος ότι είχαμε ανεπαρκές επίπεδο επενδύσεων για πολύ καιρό στην Ευρώπη. Το επίπεδο επενδύσεων ε, που χρειάζεται είναι πολύ ψηλότερο για την ενέργεια, για τις μεταφορές, για τα δίκτυα. Η Κομισιόν μιλάει για 1,3 5 τρισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2050. Και είναι τόσο, τόσο μεγάλο το ποσό που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το διαθέσει μόνη της. Θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές οι οποίες αυτή τη στιγμή βέβαια εφαρμόζουν μέτρα αυστηρής λιτότητας. Ε, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να βρούμε καινούριου τρόπους, καινούριες διεξόδους. Ένας τρόπος ε, είναι ε, νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Τα ομόλογα έργου είναι ένας τέτοιος τρόπος. Ε, πρόκειται για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έτσι ώστε να προσελκυστεί και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τον, ε, το χαρακτηρισμό της πιστοληπτικής ε, ε αξίας αυτών των ε, ομολόγων. Δεν μιλούμε βέβαια για κρατικά ομόλογα, έτσι. Είναι, και, είναι ένα ειδικός, ένας ειδικός τύπος ομολόγων. Πρόκειται για η συγκεκριμένη πρόταση αφορά 230 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2012-2013. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό για αρχή, αλλά η Κομισιόν πιστεύει ότι ε, θα μπορούσαμε ε, να ε, εξασφαλίσουμε την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ένα ποσό 20-30 φορές μεγαλύτερο με αυτή την εγγύηση. αν όλα πάνε καλά, το κόστος τελικά θα είναι μηδενικό, διότι ε, τα 230 εκατομμύρια είναι εγγύηση. Πλην όμως ε, θα πρέπει να αναλυθεί καλύτερο κίνδυνο και ελπίζουμε ότι το εργαλείο αυτό θα αναπτυχθεί πιο πολύ έτσι ώστε, όπως είπε ο κύριος Μπαρόσο, το ίδιο ανέφερε και το G20 και, η Ευρωπαϊκή, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις τελευταίες ε, μέρες και εβδομάδες. Πρέπει όμως να, να δούμε και άλλες ιδέες. Να αναλύσουμε καλύτερα την κατάσταση, έτσι ώστε να δούμε ενδεχομένω αν μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση και να αναζητήσουμε και καινούριου τύπου επενδύσεων για μικρά και μεσαία ε, project επενδύσεων, επενδυτικά σχέδια, ε, για να αυξήσουμε την, ε, ε, τη ρευστότητα στην ευρωπαϊκή αγορά, να σκεφτούμε τα ομόλογα Delors ε, ε, ομόλογα έργου ενδεχομένως τα οποία θα τα εγγυάται ο κοινοτικός προπολογισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους όσους ε, βοήθησαν, τους συναδέλφους της Επιτροπής Προπολογισμού, τον σκιώδη την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και επίσης τη Δανέζικη Προεδρία. Ελπίζουμε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα πάρει, τα, θα πάρει τη σκητάλη και θα φτάσει το θέμα αυτό στο τέλος του. Ο κύριος Μαυρογιάννης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που έχω να λάβω μέρο στη συζήτηση. Και προσβλέπω βέβαια στην ψηφοφορία πάνω στο θέμα αυτό αύριο. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονό ότι η πρόταση για μια πιλωτική φάση για την πρωτοβουλία των ομολόγων έργων μπόρεσε να προχωρήσει εγκαίρως σε κατάληξη επιτυχή. Και μπορώ ιδιαιτέρως να ε, σημειώσω με ικανοποίηση ότι αυτό ελήφθη πλήρως υπόψη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της προηγούμενης εβδομάδας. Ενθάρρυνση των επενδύσεων σε υποδομές αποτελεί κέριο στοιχείο για την υποστήριξη τη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Σε μια χρονική στιγμή όπου ασκούνται σημαντικέ πιέσει επί των εθνικών προπολογισμών, απαραίτητο είναι να κοιτάξουμε να αναζητήσουμε νέου και καινοτόμου τρόπου για να μπορέσουμε να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση λόγω τη χρηματοοικονομική κρίση γίνεται όλο και πιο ε, δύσκολη. Το οικονομικό λοιπόν περιβάλλον το οποίο αντιμετωπίζουμε μας ε, καθιστά απαραίτητο να, να δώσουμε νέες λύσεις για τις επενδύσεις στην τεχνολογία, τις πληροφορίες, τις μεταφορές, την ενέργεια. Η πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χρηματοδότηση έργων προτεραιότητας. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέσο αυτό των ομολόγων έργων μπορεί να εξασφαλίσει μόχλευση για μεγάλο όγκο επενδύσεων. Εάν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σημαντικό και με τη χρήση των ε, ομολόγων έργου θα μπορέσουμε πιστεύω να αντιμετωπίσουμε πολύ πολύ αποδοτικά και αποτελεσματικά τους λιγότερους τους πιο περιορισμένους πόρους που έχουμε. Ο όγκος αυτών των δημοσιονομικών μέσων μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον περισσότερο. Η δε συμφωνία που επιτεύχθη με το, Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντική και ευπρόσδεκτη. Ιδιαιτέρως δε, καθώς αντιμετωπίζει ζητήματα σημαντικά για το Συμβούλιο, συμβάλλει στην ε, ταχύτερη κατά το δυνατόν θέση λειτουργία αυτής της πρωτοβουλίας αναφέρεται στην κρίσιμη πρώτη φάση και την αξιολόγηση μετά την πιλωτική φάση της λειτουργίας του συστήματος έτσι να μπορέσουμε να δούμε την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες αυτού του μέσου. Πολλές από τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου ήταν κοινέ για μας. Θέλουμε ταχύτατη πρόοδο και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία της Δανίας για τον πολύ αποτελεσματικό τρόπο και αποδοτικό τρόπο με τον οποίο διεύθυνε τις επραγματεύσεις. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης για την ε, ε, δεκτικότητα και την ταχύτητα με την οποία προχώρησαν σε μια συμφωνία. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη προς τον κύριο Γκόραν Φέρμ για τον εξαίρετο τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύτηκε το τόσο σημαντικό αυτό θέμα για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τις διαπραγματεύσεις. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει περισσότερο από ό,τι ποτέ να δώσουμε όθηση σε μια ευφυή αποδοτική βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μέσα για να το καταφέρουμε και χαίρομαι ιδιαίτερω διότι σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορέσαμε εμεί από το Συμβούλιο να εξασφαλίσουμε την πρόοδο στην συμφωνία αυτή για τα ομόλογα έργου που θα συμβάλλουν σημαντικά στι επενδύσει για τι υποδομέ και ως εκ τούτου θα βοηθήσουν ε, στην ανάκαμψη της, της οικονομίας και τη δημιουργία της συνεργασίας. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω όλοι θέλουμε και επιθυμούμε. Σε ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Thank you. And now, um, I welcome also Ο λόγος στον Επίτροπο Ρέν. Uh, uh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Γκέραν Φέρμ, τους συνσηγητές Λάγκεν και Κάντσιαν και τους κοιόδης εισηγητές για τις πολύ ουσιαστικέ παρατηρήσεις τους και τα επικοδομητικά του σχόλια και προτάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον πρόεδρο τον κύριο Χόγερ για την εξαιρετική, εξαιρετική του συνεργασία κατά τη διάρκεια της ε, προετοιμασίας ε, της προπαρασκευής. Ε, να βάλουμε αυτή την πρωτοβουλία στο γενικότερο πλαίσιο της, των μέτρων ανάπτυξης ε, ε, ξεκινάμε την πρώτη φάση των ομολόγων έργου ε, ενισχύοντας την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να παρέμβει. Ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για νέους ανέργους project που τους αφορούν αυτές, οι πρωτοβουλίες είναι αυτές που αποφασίστηκαν και θα εφαρμοστούν. Χαίρομαι που η Πρωτοβουλίε που πρότεινε η Κομισιόν εδώ και αρκετό καιρό γίνονται πλέον πραγματικότητα. Και αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι κρίσιμο. Η κρίση χρέους βρίσκεται στο τρίτο έτος της. Αλλά η χρηματοπιστωτική κρίση είναι ακόμα πιο παλιά. Ο συνδυασμός αυτών των ε, δύο ε, ε, επιδεινώνει και συστημικά προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοιου είδου για να δώσουμε ένα περιθώριο αναπνοής στα κράτη-μέλη τα οποία πιο πολύ έχουν πληγεί. Την Τελευταία εβδομάδα η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης ε, αποφάσισε μέτρα που θα μας επιτρέψουν να διασπάσουμε ε, τον φαύλο κύκλο ε, που περιλαμβάνει το κρατικό χρέος και τις τράπεζες και να βελτιώσουμε την αξιοπιστία της, των οικονομιών μας. Σύντομα θα μπει σε ισχύ και ο μόνιμος μηχανισμός διάσωσης ε, που θα επιτρέψει την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών κατευθείαν χωρίς ε, δανεισμό ε, των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν προετοιμάζει την πρότασή της για τον, την, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ε, μηχανισμό επιτήρηση των τραπεζών που θα περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, αυτό θα αποτελεί τον πυρήνα της μελλοντικής ε, ενιαίας τραπεζικής, συγγνώμη, της μελλοντικής τραπεζικής ένωσης στην Ευρώπη. Προτείναμε τα σχέδια, τα ομόλογα έργου της Ευρώπης 2020 πέρσι τον Οκτώβρη ως ε, έναν τρόπο χρησιμοποίησης του βαρικού προπολογισμού ε, για μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουμε στους πολίτες και στις αγορές ότι λειτουργούν ε, μέσω αυτής της πιλωτικής φάσης που προτείνουμε. Αυτή είναι η πρόταση που ψηφίσατε ε, και που θα ψηφίσετε και σας ενθαρρύνω να την υπερψηφίσετε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη και απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χόβερ. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που συμμετέχω σε αυτήν την συζήτηση ε, σχετικά με τα ε, ομόλογα έργου. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να, ευχαριστήσω ιδιαίτερος τον εισηγητή κύριο Φέρμα, για την ρεαλιστική του προσέγγιση. Γνωρίζουμε όλοι ότι θα υπάρξουν τεράστιες επενδυτικέ ανάγκες ε, τα επόμενα έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω, αυτή η πρωτοβουλία ε, έφτασε πραγματικά στην ώρα της. Ε, υπάρχει επίγουσα ανάγκη επανεκκίνηση της οικονομίας, να σταματήσει η ολοένα ανερχόμενη ανεργία και να ξαναθετεθεί η Ευρώπη σε μια νέα θέση στον κόσμο. Μεταξύ άλλων λοιπόν ε, ε, ε, στοιχείων και εργαλείων είναι ένα καλό εργαλείο το οποίο να κινήσει τις αγορές. Ε, δεν είναι, είναι μια προσθήκη ε, στην εργαλειοθήκη που έχουμε ήδη. Ε, είναι πολλοί ηγέτες οι οποίες έχουν δεσμευτεί πλέον στην βιώσιμη ανάπτυξη και η σωστή εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα δώσει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δεν επιβάλλεται κανένα επιπλέον άχθος στους προϋπολογισμούς μέσω αυτών των project project bonds. Ε, ε, ε, τα, οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανακατευθύνονται απλώς όλα τα στοιχεία αυτά πιστεύουμε ότι θα βελτιώσουν την κατάσταση του χρέους ε, και θα οθήσουν τους επενδυτές να αγοράσουν τα ομόλογα αυτά έτσι ώστε να βοηθήσουν την κατάσταση στην Ευρώπη. Το πολλαπλασιαστικό ε, αποτέλεσμα μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και βεβαίως ε, ε, θα έχουμε την δυνατότητα να στηρίξουμε 4,3 ε, ευρώ ανά έργο σε αυτήν την περίπτωση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης και επομένως θα διατεθούν στην ουσία τελικά περαιτέρω πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ να ευχαριστήσω βεβαίως και τον Επιτροπό Όλη για την εξαίρετη συνεργασία. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορέσουν να βοηθήσουν μέσω τεχνογνωσίας ε, και μέσω πρακτικών ε, έτσι ώστε να στεφτεί από επιτυχία η κίνηση αυτή. Μέσω των κοινών εργαλείων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να απομονώσει και να ταυτοποιήσει τα προγράμματα αυτά τα οποία μπορούν να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να προωθηθούν λοιπόν οι αγορέ Ευρωπαϊκής ε, και να ε, οδηγηθούμε σε καλές και υλοποιήσιμες ε, συμφωνίες οι οποίες θα αφορούν σημαντικούς όγκους επενδύσεων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να στηρίξουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη την διαρκή πρόσβαση σε σταθερή χρηματοδότηση ε, και βεβαίως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από στήριξη έργων υποδομής είτε πρόκειται για, για σιδηροδρόμους είτε πρόκειται για άλλες υποδομές έτσι θα ανοίξουν οι προοπτικές για την Ευρώπη και ευελπιστούμε ότι τα ε, ομόλογα έργου θα ανοίξουν την όρεξη και των ιδιωτών επενδυτών έτσι ώστε να επενδύσουν περαιτέρω και σε άλλους τομείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Λάγκεν. vielen Dank, Herr Präsident. Ich... Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω να σας παρουσιάσω την γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας με 28 τροπολογίες που εγκρίθηκαν ομόφωνα. Η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών τις έκανε δεκτές ε, και τις ενσωματώνει. Ε, προκειμένου να υπογραμμίσουμε λοιπόν αυτή τη σημασία αυτή τη πιλωτική φάση. χρειάζεται μια ενδιάμεση αξιολόγηση, μια ενδιάμεση έκθεση δηλαδή, ώστε να δούμε ότι και η τεχνική αξιολόγηση βρίσκεται υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και όχι αποκλειστικά και μόνο στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε ιδιωτικό κεφάλαιο για τα μεγάλα έργα υποδομών, για την ενέργεια, για τις μεταφορές και ιδιαίτερα στην φάση της πρώτης επιλογής, ε, κύριε Χόια, θα σας παρακαλέσω να μεριμνήσετε έτσι ώστε να είναι τα καλύτερα σχέδια εκείνα τα οποία θα επιλεγούν ώστε να μην έχουμε κίνδυνο αποτυχίας. Μια πολύ αυστηρή επιλογή λοιπόν, μια πολύ αυστηρή ε, προβολή των έργων που θα ε, επιλεγούν γιατί χρειαζόμαστε αυτά ομόλογα έργου και χρειαζόμαστε και κινητοποίηση ιδιωτικού κεφαλαίου. Ευχαριστώ θερμά. Κύριος Καντσάν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εγώ είμαι απολύτως ε, υπέρ αυτής της πιλωτικής φάσης ε, των ε, ομολόγων έργων, γιατί και η αρχή χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων με την τεχνογνωσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έτσι ώστε να δημιουργηθεί η δυνατότητα υλοποίησης καλών και ποιοτικών προγραμμάτων είναι κάτι πάρα πολύ καλά. Τι δεν λειτουργεί ο προϋπολογισμός για αυτό το πολυ, ε, πρόγραμμα είναι πάρα πολύ λίγο, κυρίως αυτά τα δέκα για την ε, με τον τομέα της ενέργειας. Αυτό φαίνεται να είναι μια συμβολική κίνηση, μια συμβολική χρηματοδότηση. Θα πρέπει στο μέλλον η χρηματοδότηση να είναι σοβαρή. Ε, λείπει λοιπόν και η, η θέληση, η βούληση, το θάρρος έτσι ώστε εμείς να είμαστε αυτοί που θα πρωτοστατήσουν στην ανάκαμψη. Ε, λείπει η βούληση για την ε, πραγματική δημιουργία ενός συστήματος PPP που θα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και θα μπορέσει να σύρει την οικονομία ε, έξω από αυτήν την κατάσταση ε, την οποία, ε, στην οποία έχει βρεθεί. Δεν αναφέρομαι στο παρελθόν, ανακεφαλαιοποιήσεις, κοινή τοποθέτηση του χρέους κτλ. Αναφέρομαι στο μέλλον. Αυτό είναι ο δρόμος για γρήγορη ανάπτυξη, για δημιουργία ανταγωνιστικότητας, αυτή της ανταγωνιστικότητας που αξίζουμε δηλαδή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρικέ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς ε, να χαιρετήσω τη δουλειά του Γκόραν Φέρμα, ο οποίος ήταν πολύ παραγωγικός σε αυτό το θέμα και χάρη στη δουλειά του και τη συνεργασία με το Συμβούλιο υπό την Προεδρία της Δανίας και τώρα της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή ε, τώρα το καλοκαίρι αυτή η απόφαση. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μέσο λοιπόν, χρηματοδοτικό μέσο το οποίο καινοτομίω προς την ευφυή αξιοποίηση των περιορισμένων όπως γνωρίζουμε πόρων με βάση φυστάμενε σειρέ στον προπολογισμό αλλά και πρόσκληση νέων επενδύσεων αφετέρου. Η δημοσιονομική σταθερότητα μπορεί να φέρει ε, αποτέλεσμα μόνο με μέτρα ανάκαμψη. Ακριβώς, λοιπόν αυτά τα μέτρα που μπορούν να παραχάγουν θέσει εργασία ε, υποστηρίζουν τα ομόλογα έργου. Ιδιαίτερα για την, ε, κοινωνία, για την τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και για, τις και για την ενέργεια και τις μεταφορές. Πρέπει να προσδιοριστεί πιο συγκεκριμένα λοιπόν το έγγραφο, το μέσον, να θεσπιστούν τα μέτρα εποπτείας και να ε, να επιβεβαιώνονται οι επιτυχίες χωρίς να αποθαρρύνονται οι αγορές, να αξιοποιείται το παραγόμενο αποτέλεσμα και να αξιοποιείται το σύστημα των εγγύσεων για τις ενεργειακές επενδύσεις μαζί με τα ομόλογα έργο. Και για να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι ίσως ε, είμαστε μάρτυρες στην ανάπτυξη μιας μικτής οικονομίας, χρηματοοικονομικής ε, χρηματοπιστωτικής οικονομίας, δηλαδή και το δημόσιο τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ιδιωτικών βλέπουμε να αρχίζουν να συμπράττουν μέσα σε πολυετή έργα όπως το Connecting Europe Facility, η διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Και ευχαριστώ τώρα η κυρία Αγιάλα Σάντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι καλύτερο από άσχημα και δυσάρεστα νέα. Ε, συνεπώς θα πρέπει να ευχαριστήσουμε, να συγχαρούμε τον κύριο Φέρμ αλλά και όλους τους συνεργάτες και όλα τα θεσμικά όργανα τα οποία συνεργάστηκαν την Κομισιόν, το Συμβούλιο, ε, το Κοινοβούλιο βέβαια αυτό προφανώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που ε, ως τώρα εμφανίζεται και εξαφανίζεται και, και αναμένουμε από αυτή να είναι πάντοτε ορατή και συνεχώς παρούσα για να διαχειριστούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα λίγα δημόσια κρατικά κονδύλια που έχουμε και να τα συνδυάσουμε με ιδιωτικά κονδύλια ε, ιδιαίτερα σε αυτούς τους ε, τομείς που είναι πολύ σημαντικοί για την διακίνηση αγαθών, κυκλοφορία προσώπων, κεφαλαίων και υπηρεσιών. Ε, ε, οι υποδομές αυτές θα είναι καινοτόμες, ευφυείς, ε, θα στρέφονται προς το μέλλον και θα συνδέσουν την Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και την Ευρώπη εσωτερικά και θα δημιουργήσουν πλούτο, ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι υπάρχουν άλλες περιοχές του πλανήτη που ε, αναπτύσσονται ραχδαία. Χρειαζόμαστε λοιπόν και εμείς να παρακολουθήσουμε αυτή την ανάπτυξη ε, και νομίζω ότι αυτά τα ομόλογα θα βοηθήσουν έτσι ώστε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί ε, και ε, στην εχμή του δόρατος στους κλάδους της, ε, αυτών των υποδομών, των μεταφορών, της ενέργειας, των δικτύων κλπ. Υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση και ελπίζω ότι στα επόμενα δύο χρόνια που απομένουν για τη θητεία μας η Κομισιόν θα μας αναφέρει θετικά επιτυχή αποτελέσματα. Η ενημέρωση κάθε έξι μήνες είναι σημαντική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναμένουμε εμείς και οι πολίτες πάρα πολλά από αυτό το project. Ως συνεισηγήτρια του προγράμματος ε, συνδεδέοντας την Ευρώπη χαιρετίζω αυτό το βήμα πρόοδου προς υποδομές ευφύης ε, και βιώσιμες. Η κυρία Γιάνσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδας ALDE ε, πρέπει να σας πω ότι στηρίζουμε αυτή την, αυτή πρόταση γιατί είναι πάρα πολύ θετική. Ήταν ε, πολύ θετικό επίσης που μπορέσαμε να το ξεκινήσουμε τόσο γρήγορα. Να ευχαριστήσω βεβαίως και τον κύριο Γκόραν ε, για την εργασία του η οποία κατέληξε σε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα. Ε, δεν μας είναι στην Δανία ε, ξένη η ιδέα των υποχρεωτικών ε, δανεισμών. Με αυτό το σύστημα κάναμε ας πούμε τη γέφυρα μέχρι τη Σουηδία. Δηλαδή κάποια εταιρεία κατασκεύασε τη γέφυρα αυτή και μετά ε, πήρε τα χρήματα της πίσω μέσω των ε, συνεισφορών του κεφαλαίου. Δηλαδή εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό το σύστημα μπορεί να δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα αλλά βεβαίως γνωρίζουμε ότι ειδικά σε περιπτώσεις σαν αυτή που διανύουμε τώρα όπου τα δημόσια ταμεία δεν θα μπορέσουν για πολύ καιρό ακόμα κατά την άποψή μας να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικό. Επίσης και στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουμε δει κάτι παρόμοιο και πιστεύουμε ότι ε, με τον τρόπο αυτό σε 10 χρόνια περίπου θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ομολογιακή αγορά η οποία θα μας δώσει ενδεχομένως την δυνατότητα να στηρίζουμε από μόνοι μας ε, τα προγράμματά μας. Αυτή τη στιγμή όμως χρειαζόμαστε στήριξη. Θα πρέπει να υπάρξει, να δημιουργηθεί μάλλον το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης έτσι ώστε οι επενδυτές να πιστέψουν ε, σε αυτά τα προγράμματα, σε αυτά τα έργα και να επενδύσουν ειδικά σε αυτήν την φάση εκκίνησης. Θα πρέπει να υπάρξει καλή συνέχεια επίσης όσον αφορά τις εμπειρίες της πιλωτικής φάσης έτσι ώστε να συνεχίσουμε με καλύτερο τρόπο ε, στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει, μάλλον ε, μπλε κάρτα από τον ε, κύριο Μάρτιν. Θέλετε να δεχτείτε. Ναι βεβαίως. Κύριε Μάρτιν παρακαλώ να θέσετε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε σαν μιλήσατε για την εμπειρίες από τη Δανία. Σε αυτά τα ομόλογα έργο, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα ως προς την ανάληψη εγγυήσεων, της εγκυοδοσίας δηλαδή και δεν ανησυχείτε μήπως χρειαστεί μια εξασφάλιση εκ των στερών; Εν τέλει δε, μήπως τελικά χρειαστεί το δημόσιο να δεσμεύσει ασφαλιστικά ταμεία, στεξιδοτικά ταμεία για να δώσει εγγύησεις. Πώς θα καλυφθεί αυτό το σύστημα. Er øh, λοιπόν, είναι αυτονόητο <clears throat> ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ε, και τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να διασφαλίσουν την απαραίτητη εγγύηση για τους ε, ε, επενδυτές και για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Αλλά ξέρετε αυτό είναι μια προβληματική η οποία αφορά όλα τα ομόλογα και τα κρατικά ομόλογα δεν έχουν πολύ μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά ε, πλέον ε, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ικανοποιητικό ε, επίπεδο ασφάλειας και να υπάρχει ε, τέτοια εγγυοδοτική ας διαδικασία η οποία να επιτρέπει εις τους επενδυτές να έχουν την απαραίτητη ασφάλεια έτσι ώστε και εγώ η ίδια ή ο κύριος Μάρτιν όταν θα βγούμε στη σύνταξη τα πράγματα να είναι θετικά, να μην έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Η κυρία Ντουρό είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός, όπως είπαν και άλλοι, ότι το κράτος ε, των ε, δημοσίων οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι τέτοιο που κανένα εργαλείο δεν περισσεύει έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες επενδυτικές δυνατότητες είτε στα δίκτυα μεταφορών, είτε στην ενέργεια, είτε ε, στην, ε, ε, στην ευρυζωνική επένδυση της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα πρέπει εξ αρχής όμως να καθορίσουμε τα κριτήρια επί των οποίων θα βασιστεί η αξιολόγηση της πολιτικής φάσης. Επομένως προσοχή. Πρώτον η επιλογή των προγραμμάτων. Είναι γεγονός και ευχαριστώ εδώ τον εισηγητή ότι δουλέψαμε για τα κριτήρια, τα πολύ σημαντικά κριτήρια διάρκειας στην φάση της επιλογής γιατί όλα ε, τα, ε, ε, όλα τα προγράμματα δεν είναι το ίδιο καλά για την Ευρώπη. Επομένω, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την ποιότητα. Δεύτερον, το θέμα των κινδύνων. Βεβαίω, αντικειμενικά υπάρχει ένα οικονομικό κίνδυνο, βεβαίω μπορούμε να τον ελαχιστοποιήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά υφίσταται. κατά αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στη φάση τη αξιολόγηση, δηλαδή να δούμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα μα επιτρέψουν να μειώσουμε ε, στο λιγότερο δυνατό τον κίνδυνο. Εγγυόμενοι βεβαίω βεβαίω ε, και τι ε, επενδύσεις και τι δάξεις κτλ. Ε, βεβαίω πρέπει να ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά οπωσδήποτε εξ αρχής να καθοριστούν τα κριτήρια πριν περάσουμε στην γενικοποίηση αυτού του έργου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο είναι απαραίτητο βεβαίω, αλλά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αντιμετώπιση του εδώ τώρα στην αρχή του. Ευχαριστώ πολύ χαιρετίζω τις προτάσεις του εισηγητή, ιδιαίτερα για τις επενδύσεις που θα βοηθήσουν ε, να ε, ε, δώσουμε όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά θα πρέπει να είναι επενδύσεις με πραγματική αξία. Διασυνοριακή σύνδεση δικτύων μεταφορών, ενέργειας, ευρυζωνικών υπηρεσιών, πραγματικά επενδύσεις με ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Παλιότερα επενδύσεις σε υποδομές δεν είχαν τέτοιου είδους αξία πάντοτε. Ε, επίσης, συμφωνώ με την προσέγγιση ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Πρόκειται όμως για ένα πιλωτικό σχέδιο, συνεπώς έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Στο τέλος αυτής της περίοδου ε, θα τεθεί υπό ανεξάρτητη ανάλυση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι επίσης σημαντικό η ανάλυση αυτή να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Γιατί δεν θα πρέπει να είναι απλώς εθιμοτυπική ή τυπική ε, το κλειδί θα πρέπει να είναι η προστασία των συμφερόντων και της έκθεσης των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Ο, η, η κύριος Ενά. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, πρέπει να δώσει στην Ευρώπη υποδομές. Πολύ καλό αυτό. Και θα ήταν ακόμα καλύτερο αν κατέληγε σε μια κρατική ε, ιδιοκτησία αυτών των υποδομών. Δηλαδή, αν καταλήγαμε σε δημιουργία κρατικών δικτύων μεταφοράς ενέργειας, ευρυζωνικών υπηρεσιών κλπ. Θα πρέπει να ε, ε, τελειώνουμε με μια ανταγωνιστικότητα με τον ιδιωτικό τομέα που οδηγεί σε ανισότητες, σε διαφθορά, σε πολύ υψηλές τιμές για τη χρήση των υποδομών κλπ. Χάρη στο δόγμα του ανταγωνισμού έχουμε φορτηγά τα οποία κινούνται στην Ευρώπη κενά και καταναλώνουν πιο πολύ ενέργεια από ότι αυτήν που μεταφέρουν. Αν η Ευρώπη θέλει να μπει στον 21ο αιώνα και να μην επιστρέψει στο 19ο, θα πρέπει να πει όχι στον στήρο ανταγωνισμό και ναι στην συνεργασία και τη συμπληρωματικότητα. Το σύστημα χρηματοδότησης αυτών των υποδομών είναι απαραίτητο αλλά δεν θα πρέπει να υποβοηθούμε επιχειρήσεις ε, ενεργειακές οι οποίες μας οδηγούν σε αδιέξοδο. Εγώ έχω να σας προτείνω μια καινοτόμα λύση που είναι σύμφωνη με το διεθνές συμφέρον, συμφέρον των ευρωπαϊκών πολιτών. Θα πρέπει να γίνει, να γίνει χρηματοδότηση αυτών των υποδομών με τον ίδιο τρόπο, κρατικό και ευρωπαϊκό, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η αναχρηματοδότηση, η ανακεφαλαιοποίηση των ε, τραπεζών αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Μοργάντη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετική η πρόταση αυτών των project bonds ε, έτσι ώστε να αναπτυχθούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας. Τα 230 εκατομμύρια ευρώ βέβαια δεν είναι ικανή χρηματοδότηση σε σχέση με την πραγματική ανάγκη όμως. Ε, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πρόκειται για μια πρώτη πιλωτική φάση και παρά ε, την έλλειψη όσον αφορά τη χρηματοδότηση θεωρώ ότι τα επιτευχθέντα είναι ήδη πάρα πολύ σημαντικά. Εν πάση περιπτώσει είναι χρήσιμη η διαδικασία αυτή έτσι ώστε ε, να καταλάβουμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης ε, επενδύσεων όσον αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια και την επικοινωνία στην Ευρώπη. Ελπίζω πάντως ότι τα προγράμματα που θα συμμετέχουν σε αυτήν την πιλωτική φάση θα έχουν επιλεγεί με μεγάλη προσοχή και ότι στο τέλος της πιλωτική φάσης ε, θα γίνει μια πολύ προσεκτική αξιολόγηση. Δεν μπορούμε να επενδύουμε ε, δημόσιο χρήμα σε ε, επικίνδυνες επενδύσεις με επισφαλές αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σόζα Βάγκνερ. Συνάδελφοι, εστιάζουμε την προσοχή μας στις ε, τράπεζες ε, από τις οποίες για τις οποίες ε, επανειλημμένως ακούμε ότι είναι το αίμα του κοινωνικού ιστού. πολύ ωραία. Κάθε σώμα όμως έχει αρθρώσεις και σπονδυλική στήλη. σπονδυλική στήλη και οι αρθρώσεις του κοινωνικού σώματος το οποίο ονομάζουμε Ευρώπη είναι τα δίκτυα μεταφορών και τα δίκτυα υποδομών, ενεργειακών υποδομών. Είναι απαραίτητο να κινητοποιήσουμε την ιδιωτική χρηματοδότηση και στην συγκεκριμένη περίπτωση και την κρατική χρηματοδότηση. Είναι και ευκαιρία ταυτόχρονα για να ε, προωθήσουμε την έκδοση ιδιωτικού χρέους ε, με εγγύηση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρήση σε, αυτούς τους, σε αυτές τις υποδομές και θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλους τους επενδυτές. Συγχαρητήρια για την εργασία του εισηγητή και των συνεισηγητών και στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Πολέδο. Γκαρίγα Πολέδο. Ε, προσωπώ τους ε, σοσιαλιστές στον προϋπολογισμό αλλά είμαι και ε, βουλευτής ε, που ε, εργάζεται για κοινωνικά θέματα. βρισκόμαστε σε μια περίοδο σημαντικής λιτότητας και περικοπών. Η χρήση τέτοιων κοινοτόμων χρήματο πιστοτικών εργαλείων, χρηματοοικονομικών εργαλείων είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, το, την χρονιά το Κοινοβούλιο ε, συμφώνησε για την ανάγκη εισαγωγή τέτοιων νέων εργαλείων για να αντισταθμίσει την ενδεχόμενη ανεπάρκεια του προπολογισμού. Οι επενδύσει ε, στι μεταφορέ, την ενέργεια και τι τηλεπικοινωνίε είναι απαραίτητε και πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Οι ανάγκε είναι περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ ε, μέχρι το 2020. Λαμβάνοντα υπόψη το πόσο δύσκολο είναι να εξασφαλίσει κανεί ιδιωτικό επενδυτή για μεγάλα σχέδια υποδομών, προγράμματα υποδομών, ε, η πιλωτική φάση των ομολόγων ε, έργου είναι ακόμη πιο σημαντική το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε την ε, ε, μελλοντική χρήση ε, των ομολόγων αυτών και τη σύνδεσή τους με την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Είναι ένα project πραγματικά ευρωπαϊκό, αυθεντικά ευρωπαϊκό, που προσελκύει και ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα ευρωπαϊκής αξίας. Είναι σημαντικό που σε δύο τριμερείς διαλόγους οι προτάσεις του εισηγητή έγιναν δεκτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι που θα οδηγήσει σε ε, έγκριση ε, του ε, σχεδίου σε πρώτη ανάγνωση, έτσι ώστε να εφαρμοστεί αμέσως. Είναι σημαντικό να απαιτήσουμε από την Κομισιόν να μας υποβάλει την ενδιάμεση έκθεση στο μέσο του 2013, οπότε αν οι αγορές δεν έχουν ανταποκριθεί θετικά στα ομόλογα έργου να είμαστε σε θέση να τα βελτιώσουμε για να εφαρμοστούν καλύτερα στο δεύτερο εξάμεινο του 2013. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σαλκαντράουε. Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους όσοι συνέπραξαν στο θέμα αυτό. Έχουμε συζητήσει πολύ το θέμα, το έχουμε ακούσει και από τις ειδήσει αυτό το νέο σύστημα με ομόλογα έργου που θα πρέπει να ενισχυθεί διότι μπορεί να μας φέρει πολλές ε, νέες επενδύσεις οι οποίες και άμεσα αλλά και μέσα θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύω λοιπόν ότι αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την, ε, ε τους στόχους μας θα πρέπει να βρούμε ένα μέσο χρηματοδότησης μεταξύ των, διαφόρων νέων επιλογών που θα έχουμε θα είναι και αυτά. Βεβαίως πρέπει να αποδεσμεύσουμε τα 230 δισεκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται για τη χρηματοδότηση δύο-τριών έργων. Γιατί ξέρουμε ότι σακούλι το σακούλι γεμίζει φασούλι, το φασούλι γεμίζει το σακούλι και έτσι μπορούμε να περιμένουμε ότι από τα λίγα αυτά ε, ποσά μπορούμε να διαθέσουμε αρχικά μπορούμε να έχουμε πολύ σημαντικά έργα. Τα καινοτόμα αυτά έργα μπορούν να αποτελέσουν ε, μια λύση αλλά όχι άλοθη ώστε να μην αποδεσμευθούν επενδύσεις, ποσά για επενδύσεις. Οι πιστώσεις αυτές λοιπόν για τις επενδύσεις και ιδιαίτερα για, ε, για τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη θα πρέπει να δοθούν ώστε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάλεαν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με χαρά σημειώνω ότι η ανάπτυξη είναι πλέον στο επίκεντρο των συζητήσεων. Την ανάπτυξη όμως πρέπει να τη δημιουργήσουν οι αγορές και όχι οι νομοθεσίες, όχι οι νομοθέτες. Άρα θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις αγορές αν θέλουμε ανάπτυξη. Θα πρέπει να επιταχύνουμε την ολοκλήρωση των υποδομών για να βελτιώσουμε τις συνθήκες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας. συχνά λοιπόν ε, δημοσιονομικά μας ε, μέσα θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις ε, υποδομές αυτές. Με τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη μπορούμε να έχουμε αξιοποίηση αυτών των δημοσιονομικών μέσων για πιο ουσιαστικές υποδομές μέσα σε, μια, σε ένα πλαίσιο διαφανές, σε ένα πλαίσιο αποδοτικό το οποίο δεν θα στρεβλώνει τις αγοράες και θα προσελκύει επενδυτές και δεν θα τους ε, εκδιώχνει ιδρύοντας αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Χρειαζόμαστε το ομόλογα έργου, ναι, χρειάζεται να τα αξιολογήσουμε μάλιστα και να τα βελτιώσουμε τα μια πρώτη πιλωτική φάση. Επίσης χρειάζεται να υποστηρίξουν το θεσμικά όργανα, τους εμπλεκόμενους φορείς, τράπεζες, θεσμικούς επενδυτές για να αναπτύξουν περισσότερο αυτή την νέα τάξη επενδύσεων ώστε να αποδεσμευθεί από τις, ε, τους περιττούς δεσμούς ε, και τη γραφειοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μόχλευση για κάθε ευρώ που θα δαπανά ο δημόσιο τομέα. Υπάρχει ανάγκη να δράσουμε ταχύτατα. Πια δεν έχει, δεν έχει, έχει παρέλθει πλέον η εποχή που μπορούσε μόνο με επιχορηγήσει να κάνουμε τα έργα. Ο κύριο Τουρμέ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Χόια. Πιστεύω ότι σε αυτή την ε, πιλωτική φάση είναι πολύ σημαντικά τα, περιβαλλοντικά κριτήρια γιατί θα πρέπει να σταματήσουμε να δημιουργούμε υποδομές οι οποίες μας απομακρύνουν ακόμη περισσότερο από τους περιβαλλοντικούς και τους ενεργειακούς μας στόχους ένα σημαντικό στοιχείο αδυναμίας το οποίο επισημαίνω είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί τώρα και μετά βέβαια και στο Ταμείο και στη Διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη λύσεις για ανανεώσιμα έργα, για ε, την ε, λύση που θα δοθεί ε, σε περίπτωση που αξιολογηθούν αρνητικά κάποια έργα. Η η δανική δηλαδή ενεργειακή επιχείρηση, έχει πωλήσει ένα μερίδιο από τα ανανεώσιμα σχέδιά της τα οποία μπορούν σε πρώτη φάση να θεσπίσουν και να σχεδιάσουν οι ειδικοί και στη συνέχεια ε, όπως μπορούμε να κάνουμε γενικότερα πιστεύω, να μπορούμε να προσελκύουμε επενδυτές, ιδιώτες, ε, όταν αρχίζει να αποδίδει ένα έργο. Δηλαδή ξεκινάει ο δημόσιο τομέα και στη συνέχεια το πολύ και το αναπτύσσει περαιτέρω για τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το ε, αναζητήσουμε ω λύση και ω μέθοδο για να προσελκύσουμε περισσότερα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η έκθεση την οποία ε, εξετάζομαι συστήνει ένα όργανο ε, το οποίο ε, θέλει να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα ε, ομολόγων ε, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά. Εγώ είμαι μάλλον συγκρατημένος και επιφυλακτικός. Πιστεύω ότι τα κράτη ήδη έχουν χρεωθεί αρκετά. Έχουν μεγάλο χρέος ήδη και αναρωτιέμαι αν μπορούμε να τους ε, βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή στην ουσία προσπαθώντας να βοηθήσουμε τις χώρες θα τις χρεώσουμε ακόμα περισσότερο. Δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ε, ε, επίσης στο κείμενο αναφέρεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Δεν καταλαβαίνω πώς, δεν μπορώ να καταλάβω πώς διασυνδέονται τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας με τις κλιματικές αλλαγές. Νομίζω ότι υπερβαίνει το πλαίσιο η αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μάρτιν. Έχετε τον λόγο κύριε Μάρτιν. Πρόεδρε, είναι πολύ ευφύητα όσα μας είπε ο κύριος Τουρμές και μακάρι να μπορούσε να πειράσει περισσότερο την ευρωπαϊκή πολιτική. Θα ήθελα να προσθέσω βεβαίως ότι βεβαίως ε, είναι κάπως ε, ταπεινό το πεδίο στο οποίο αναπτύσσονται αυτά τα ομόλογα έργου και η σχετική δανειοδότηση, αλλά μπορούν να δώσουν πολύ μεγάλη απόδοση. Βεβαίω, ο κίνδυνος είναι αυτός των εγγύησεων. Συγκεκριμένα, 380.000 χιλιόμετρα ε, καλωδίων για ε, διασύνδεση τεχνολογία επικοινωνιών έχουμε στη Γερμανία, ενώ θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον το πενταπλάσιο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε μεθόδους οι οποίες να είναι διάδρομοι, όχι μόνο αυτοκινητόδρομοι, όχι μόνο ε, δίκτυα ευρέως φάσματος, αλλά συνδυασμένες υποδομές που να βελτιώνουν γενικότερα την επικοινωνία της μεταφοράς και την ενέργεια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας, τον κύριο Φέρμ, για τις τεράστιες προσπάθειες του και, για, και να ευχαριστήσω και την Κομισιόν γιατί ε, άκουσε τις ε, προτάσεις ε, και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τις είχε ζητήσει να υποβάλει αυτή την πρόταση για τα ομόλογα έργο. Η Ατζέντα Ευρώπη 2020 έχει θέσει ψηλά τον πύχη και γι' αυτό το λόγο τα έργα υποδομών είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Μόνο με αυτά θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2020. Πολλά από τα υπάρχοντα δίκτυα είναι ήδη ξεπερασμένα, απερχιωμένα. Η ενεργειακή υποδομή δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως κλπ. κλπ. Θα χρειαστούν τεράστιες επενδύσεις, οποίες προφανώς δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μόνο με κρατικά κονδύλια. Βασιζόμαστε στη ε, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το τρέχον οικονομικό κλίμα, το οποίο προφανώς δεν ελκύει εύκολα ιδιωτικές επενδύσεις. Το πιλωτικό πρόγραμμα προβλέπει ένα σχετικά χαμηλό ποσό 230 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει όμως να περιμένουμε να δούμε το θετικό αντίκτυπο πρώτα που θα προκαλέσει στον ιδιωτικό τομέα και μετά να αναθεωρήσουμε το ποσό για το μέλλον. Νομίζω ότι ήδη αυτό το ποσό θα δώσει σημαντικά κίνητρα για την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ε, δικτύων υποδομών, ιδιαίτερα για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, που, ο ευρωπαϊκός προπολογισμός δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει. Κύριε Μάν, Μάναρ. Α, με συγχωρείτε, είχα ξεχάσει τον κύριο Ντεμπάκερ. Κύριε Πρόεδρε, τα ευρωπαϊκά μας δίκτυα των μεταφορών δεν είναι πλήρη, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι απαραίτητο ωστόσο στο προσεχές μέλλον μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων και της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε έργα υποδομών. Αυτέ ο δανεισμός μέσω των ομολογικών ομολόγων είναι πολύ σημαντικός γιατί μας επιτρέπει σε περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσχέρειας να βρίσκουμε, ε, να αντλούμε κονδύλια για τις επενδύσεις και βέβαια και, κονδύλια τα οποία βρίσκονται σε ελανθάνουσα κατάσταση και τα οποία μπορούμε να ε, αφυπνίσουμε όπω είπε. Τα 230 εκατομμύρια ε, αποτελούν μόνο μια μικρή αρχή, όμως μπορούν να επιτρέψουν τη χρηματοδότηση πολλών έργων και την αντιμετώπιση ζητημάτων τεχνικής διαχείρισης για, τις, ε, ε, για τους επενδυτές έτσι ώστε στο μέλλον να μπορούμε να επενδύουμε πλήρως ε, μέσω αυτών των ομολόγων. Η ομάδα μου υποστηρίζει πλήρως την ιδέα αυτή. Ευχαριστώ κυρία Μάνερ, χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Το έχουμε πει επανειλημμένως, είναι σημαντικό η Ευρώπη να συνεισφέρει στην δημιουργία μιας λειτουργούσας υποδομής. Μόνο έτσι θα πετύχουμε οικονομικά. Στο, μέτρο, στο μέλλον θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ακόμα περισσότερο κρατικά και ιδιωτικά κονδύλια για τα ίδια project. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει όλες τις ε, υπάρχουσες δυνατότητες. Έχουμε την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, έχουμε ταμεία όπως το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν πλήρω περισσότερο από σήμερα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Επίσης, είναι σημαντικό να δούμε την Ευρώπη στο σύνολό της, να δούμε τις υποδομές της σε όλη την Ευρώπη. Να μην εστιάζουμε μόνο στο κέντρο, να δούμε και την Ευρώπη του Βορρά. Thank you. <clears throat> Now we've Σα ευχαριστώ και τώρα διαδικασία Καριστιάη με την κυρία Αντζελίλη πρώτη ομιλήτρια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εκκίνηση των ομολόγων έργου είναι μια πρώτη σημαντική φάση του Συμφώνου για την Ανάπτυξη. Πρόκειται βέβαια για ένα πιλωτικό σχήμα, το οποίο ίσως να είναι και υπερβολικά επιφυλακτικό στη λειτουργία του, αλλά παρόλα αυτά για 27 κράτη-μέλη 5 δις παραμένει συμβολικό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα συγκεκριμένο μήνυμα, συγκεκριμένο επαναλαμβάνω έτσι ώστε να προκαλέσουμε και την είσοδο ιδιωτικών επενδύσεων στρατηγικής φύσεως για να καταστήσουμε ανταγωνιστική την ευρωπαϊκή οικονομία και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Θα συμφωνήσω με αυτούς οι οποίοι υποστήριξαν ότι θα πρέπει να υπάρξει αυστηρή πειθαρχία σε σχέση με την αξιολόγηση, την αξιοπιστία των προγραμμάτων και την προσμέτρηση το σωστή ε, σε επίπεδο μεγέθους των αποτελεσμάτων. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για μια στρατηγική αυθεντική φάση ανάπτυξης για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριο Σκοφεράτη. Grazie Presidente. Abbiamo sentito questa mattina come il Presidente cipriota faccia affidamento sulla costruzione delle reti, sia quelle che riguardano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 Ευχαριστώ κύριε Σκοσλόφσκι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φάρμα, ο οποίο συνέταξε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και συμφωνώ ότι οι πολυτροπικοί διάδρομοι για τις μεταφορές έχουν κέρια σημασία αν θέλουμε να έχουμε επαφές με άλλες χώρες. Έχουμε υψηλό κόστο στι επενδύσει μα για τι ενεργειακέ γραμμέ, επί παραδείγματο. Και ω εκ τούτου χρειάζεται να εξασφαλίσουμε περισσότερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα που θα μα ε, εγγυηθεί την επιτυχία. Για τα ομόλογα έργου. Είναι πολύ σημαντικό μέσον, πρέπει να λύσουμε περαιτέρω. Είμαι βεβαίως ε, ότι τα, η πιλωτική αυτή φάση θα μας δώσει πολύ πιο συγκεκριμένη εικόνα για την ε, για το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα για το μέσον αυτό και ελπίζω επίσης ότι οι νέες δυνατότητες για επενδύσεις θα λιάνουν τις ε, διαφορές και δυσαναλογίες που επικρατούν μεταξύ διαφορετικών περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό βέβαια στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίκα. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Μια πρώτη πιλωτική φάση για τα ομόλογα έργου πρέπει να ξεκινήσει για να μπορέσουμε να δούμε την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη να λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Πρέπει το 2012-2013 να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση με εξασφάλιση χρηματοδότησης ε, και ποσά προερχόμενα από άλλα έργα. Με την πρωτοβουλία αυτή μπορούμε να αντλήσουμε μέχρι 200 ε, εκατομμύρια ευρώ από τον ε, προπολογισμό ε, για τα ευρωπαϊκά δίκτυα για τις μεταφορές και άλλα 10 για, τις, για την ενέργεια. Μπορούμε λοιπόν να διεκδικήσουμε κονδύλια με βάση έργα, προτινόμενα έργα, που μπορούν ευχερός να υλοποιηθούν. Τα κράτη-μέλη μπορούν τις ε, προτάσεις να τις καταθέσουν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2013 και μόνο σε περίπτωση περίπλοκων έργων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2014 και μπορούμε να περιμένουμε καλή απορρόφηση κονδυλίων στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ και ως Πάσκα. Πρόεδρε, Επίτροπε, ε, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται ε, ε, μια όθηση για να ξεφύγει από την ε, στασιμότητα. Η χρηματοδότηση ουσιαστικών έργων υποδομών θα βοηθήσει στην γρήγορη εφαρμογή τους και στην εξασφάλιση οικονομικής πρόοδου. Αυτό συνδέεται με την καλή χρήση τέτοιων μηχανισμών η πιλωτική φάση θα μας ε, επιτρέψει να αξιολογήσουμε το εργαλείο αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μαζί με την Κομισιόν θα πρέπει να συνεργαστούν με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι το σύστημα αυτό θα είναι βιώσιμο και αποτελεσματικό ε, ενώ θα χαρακτηρίζεται από τους ελάχιστους νετούς κινδύνους. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για να μας ε, βοηθήσει ε, να ε, υλοποιήσουμε τέτοιους project. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή τη φάση διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν κίνητρα για τις επενδύσεις στον τομέα των υποδομών στις μεταφορές, στην ενέργεια, στην πληροφορική, στις τηλεπικοινωνίες γενικότερα. Η έκδοση των ομολόγων έργου ε, θα κινητοποιήσει και περισσότερους πόρους και από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή οικονομία να επανεκκινήσει χρησιμοποιώντας αυτό το νέο μέσο με το οποίο θα πρέπει φυσικά να το γνωρίσουμε καλύτερα. Χάρη στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τα ομόλογα αυτά θα γίνουν πιο ασφαλή, θα μειωθούν οι κίνδυνοι και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ήδη σε αυτή τη φάση να φτάσουμε μέχρι 8,8 δις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λέει ο κύριος Χόιερ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την πρωτοβουλία αυτή και για τη δυνατότητα την οποία ανοίγεται στην τράπεζά μας να ε, πάρει μέρος στην εφαρμογή της συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, αρχίζουμε δουλειά με την απαιτούμενη προσοχή, ελπίζω να πετύχουμε τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα φυσικά αυτά θα αντιμετωπιστούν, θα αξιολογηθούν και θα κριθούν με αντικειμενικό τρόπο στα πλαίσια μιας ειλικρινούς προσπάθειας αξιολόγησης του ότι έχουμε πετύχει σε ένα κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι η αξιολόγηση βασικό συστατικό της επιτυχίας του μέσου αυτού και η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει επί τη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτό θα δείξει την επιτυχία ή όχι. Ένα από τα πλεονεκτήματα της τράπεζάς μας είναι ότι δεν είμαστε μόνο μία απλή τράπεζα και έχουμε το απαιτούμενο πιστοτικό προσωπικό, αλλά είμαστε και ένας οργανισμός ο οποίος έχει βαθύτατη εμπειρογνωμοσύνη στην επιστήμη της μηχανικής και γενικότερα στις θετικές επιστήμες. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί αν θέλουμε να εφαρμόσουμε σωστά τις αρχές μας, να είμαστε πιστοί στις αρχές μας και να ελέγξουμε σωστά τα προγράμματα και σε επίπεδο τεχνολογίας και σε επίπεδο τεχνικής βιωσιμότητας και σε επίπεδο οικονομικό, απαιτείται αυτή η εμπειρογνωμοσύνη που θα δώσει εγγυήσεις στην διαδικασία. Φυσικά έχει δίκιο όταν λέει το ε, σχέδιο των ομολόγων έργου εγγυήσεων η χρηματοδότηση της ενεργειακής παραγωγής έτσι δεν είναι εφικτή και εγώ θλίβομαι γι' αυτό εν μέρη. Θα πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε αν στο μέλλον ο προγραμματισμός αυτών των δυνατοτήτων και άλλων διαθροτικών κονδυλίων μπορεί να αναδιοργανωθεί, να δρούμε ταχύτερα θα μπορούσαμε να δρούσαμε ταχύτερα σε σχέση με κάποιες δραστηριότητες. Αυτό θα είναι μια ευκαιρία που σε συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής Συμβουλίου και από κοινού με την Τράπεζα θα πρέπει να δράσουμε. Θα είναι ενεργή, ενεργός η Τράπεζα ε, και στο μέλλον και σε σχέση και με τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική και αλλού και κανένας δεν θα ξεπεράσει τις προσπάθειές μας. Τελευταία παρατήρηση για τον κίνδυνο, δύο λόγια. Κυρίες και κύριοι, φυσικά υπό τις συγκεκριμένες αυτές πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα εγγυάται μόνο το 20% του ε, παλαιού αυτού χρέους και δεν θα έχουμε το θέμα των ε, ομόλογων και θα έχουμε και ένα μερίδιο, ένα ε, μέρισμα σε σχέση με τα όσα θα παρέχουμε γιατί σε σχέση με την 100% ε, εγγύηση που δεν είναι δεδομένη υπάρχει ο κίνδυνος στην αγορά και θα πρέπει εδώ να επιλέγονται τα πιο υγιή σχέδια και θα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός για την λήψη αποφάσεων. Αυτό θα έχει σημασία κλειδιού για τις αποφάσεις μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέν παρακαλώ τώρα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Μπορώ και εγώ να προσθέσω την φωνή μου στα σχόλια του Πρόεδρου και ευχαριστώ για μια ουσιώδη και επικοδομητική συζήτηση. Και επίση θέλω να σας ευχαριστήσω για την στεναρή υποστήριξή σας για το σχέδιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 για τα ομόλογα έργου και για τα κίνητρα που θα δίνονται στις ιδιωτικές επενδύσεις μέσω κοινή ανάληψης ε, κινδύνων μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να χρησιμοποιηθούν σε μια ευρύτερη κλίμακα προσπάθεια στις υποδομές. Είναι σημαντικό να εξειδικεύσουμε αυτά εφόσον θα έχουν εγκριθεί από πλευρά σας οι προτάσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα προσυπογράψουν μια συμφωνία συνεργασία όσο το δυνατόν γοργότερα μετά από την έγκριση αυτής της πρότασης τελικά από το Συμβούλιο τον Ιούλιο όπως αναμένεται. Και όσον αφορά εξειδικευμένα συγκεκριμένα σχέδια, από ό,τι γνωρίζω η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήδη ε, λαμβάνει ε, προσφορές από ενδιαφερόμενους ε, για τέτοιου είδους πιθανά σχέδια για τους διαφορετικούς τομείς μεταφορών, για παράδειγμα ενεργειακού τομέα και τηλεπικοινωνιών για να, ξεκινήσουν, ε, να, να ξεκινήσει η διαδικασία υπογραφών και έγκριση στο δυνατόν γοργότερο. Φυσικά γνωρίζουμε ότι η πιλωτική αυτή φάση έχει ένα προϋπολογισμό 230 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά μόνον. Αυτό τι σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πιλωτική φάση ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε να εξευρεθεί αυξημένη ε, δυνατότητα επενδύσεων για αυτά τα σχέδια στο μέλλον και για τις τηλεπικοινωνίες και για τις ε, ε, μεταφορές και για την ενέργεια και για την πράσινη ανάπτυξη συνολικά. Και πραγματικά σε αυτή την πιλωτική φάση θα πρέπει να λιάνουμε, να προλιάνουμε το έδαφος ώστε να υπάρξουν ενδυναμωμένες, ενισχυμένες παρεμβάσεις από πλευράς του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ευδοκιμήσουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Αυτά τα ομολογά τα θεωρούμε ως έναν απόσπαστο σημαντικό τμήμα ώστε να μπορέσουμε από το 2014 και εφεξής να δράσουμε αποτελεσματικά. Σημαντικό παράδειγμα για την δράση μας για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, οι δεσμεύσεις από πλευράς των νέων κρατών μελών και της Ένωση συνολικά για να αντιμετωπιστεί η σημερινή κρίση και να κινητοποιηθούμε ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και η ανάπτυξη είναι σημαντικότατες υποθέσεις και πρέπει έτσι να αντιμετωπίζονται διότι η ευημερία κάθε Ευρωπαίου πολίτη εξαρτάται από την ευημερία της Ευρώπης συνολικά στο επίκεντρο δυσχερών εθνικών συζητήσεων είναι αναγκαία αυτά τα πολιτικά μέτρα και εξετάζοντας αυτά έχει κέρια σημασία να μπορέσουμε να καταδείξουμε τα ωφέλη της Ευρώπης και αυτής της δράσης με συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα υπέρ των πολιτών και να το κάνουμε, να το πράξουμε αυτό αποτελεσματικά το δυνατόν ταχύτερα. Ένας επιπλέον λόγος αυτός γιατί τα ομόλογα έργου διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο για την συνολική προσπάθεια υπέρ της ανάπτυξης από την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Τέλος ο κύριος Φέμ. Α, με συγχωρείτε, κύριος Μαυρογιάννης. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτές. σεβόμενος ε, ορισμένες ε, διαφοροποιούμενες απόψεις πιστεύω ότι είναι μία από τις σπάνιες στιγμές που έχουμε εξαιρετικά ευρία πλειοψηφία για καινοτόμες ιδέες και σας ευχαριστώ όλους για την πολύ οικονομική συζήτηση. Ορισμένοι είπαν ότι τα 230 εκατομμύρια ε, είναι χαμηλό ποσό αρκετά χαμηλό. Αλλά ευθύ εξ αρχή είπα ότι αυτό το ποσό θα πρέπει να παίξει ρόλο μοχλού για πολύ μεγαλύτερε επενδύσει στο μέλλον. Πολλοί τόνισαν την ανάγκη να επιλεγούν προσεκτικά τα προγράμματα. Σύμφωνο πολύ. Πρέπει επίσης ε, να διασφαλίσουμε ότι μακροπρόθεσμα θα προστίθεται αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι και ο πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως και ο Επίτροπος Ρεν έδωσαν τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις ε, σε σχέση με τα θέματα αυτά συμφωνώ επίσης με εκείνους που τόνισαν την σημασία της ε, εκτίμησης. Τα επόμενα βήματα θα είναι κλειδί. Μόλις το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εγκρίνουν το κείμενο, θα ξεκινήσει η εφαρμογή των πιλωτικών προγραμμάτων, θα υπάρξει χρηματοδότηση προγραμμάτων και θα αποτιμήσουμε πώς ε, θα γίνει δεκτή αυτή η πρωτοβουλία από τους ε, παράγοντες της αγοράς. Η Επιτροπή και η Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να διατηρήσουν έναν ε, στενό διάλογο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Σε αυτά τα πρώτα βήματα ούτω ώστε να εξαχθούν τα σωστά διδάγματα από την πιλωτική φάση για να ληφθούν υπόψη για την δεύτερη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, ο κύριος Φέρμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτήν τη διαφωτιστική συζήτηση. Ε, λίγα σχόλια, καταληκτικά. Πρώτον, την ανάγκη του μέσου αυτού. Ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ευρώπη είναι οι ανεπαρκείς επενδύσεις και δεν είναι κάτι το προσωρινό αλλά διαρθρωτικό. Η σημερινή κρίση όμως ε, κάνει την κατάσταση αυτή πολύ πιο δυσκίνητη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε νέα συμπληρωματικά μέσα. Τι προγράμματα θα χρηματοδοτήσουμε. Συμφωνώ με τον κύριο Χόιερ. Ε, θα επικεντρωθούμε στις πιο αναπτυσσόμενες αγορές, αλλά ευχαριστώ τον πρόεδρο Χόιερ που τόνισε ότι ίσως είναι δυνατή μια ευρύτερη προοπτική στο μέλλον το μέσο αυτό να μπορεί να ε, αφιερωθεί και σε άλλους στόχους. Για τα κριτήρια, ο κύριος Τούρμας και μερικοί άλλοι έθιξαν ε, την ιδέα και άλλου τύπου προγράμματα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βεβαίως, ε, θετικά το αντιμετωπίζουμε. Το συζητήσουμε στα πλαίσια του προσεχούς ε, ε, δημοσιονομικού πλαισίου, στα πλαίσια των προγραμμάτων έργου. Πολύ ανοιχτά το βλέπω η κύρια συζήτηση ε, αφορούσε τον κίνδυνο. Ξέρω ότι κάποια κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου, είναι απρόθυμα να αποδεχτούν αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά ελπίζω ότι η συζήτηση έχει μειώσει τι ε, ανησυχίε του. Δεν θα διατρέξουμε με τα χρήματα των φορολογουμένων ε, παράλογου κινδύνου. Χρειαζόμαστε αυτή την επιπλέον προσπάθεια. Κοινωνικοποιούμε του κινδύνου και ιδιωτικοποιούμε τα κέρδη. Με τι εγγυήσει που συζητήσαμε μπορούμε να κινητοποιήσουμε πόρου που αλλιώ θα έμεναν στα χρηματοκιβώτια ή θα περνούσαν στην κερδοσκοπία, αυτοί που θα κερδίσουν περισσότερο θα είναι φυσικά φορολογούμενοι. Ο κίνδυνος νομίζω ότι είναι αυστηρά περιορισμένος. Δεν θα υπάρχουν ε, ε, ιδιαίτεροι κίνδυνοι και αν δώσουμε 230 για επενδύσεις ή μάλλον συγγνώμη, για ε, ε επιδοτήσεις που θα οδηγήσουν σε άλλα 230 εκατομμύρια επενδύσεις τότε θα τα έχουμε πάει καλά. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή Προπολογισμών. Η γραμματεία της έκανε θαυμάσια ε, εργασία και όπως επίσης και οι δικοί μου συνεργάτες και τους οποίους ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φέρμ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Χόε και κύριε Μαυρογιάννη. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Λίγη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Και τώρα.